make a start on the explanations of vote. Για να αρχίσουμε με τις επεξηγήσεις δηλώσεις πρώτα-πρώτα όσον αφορά την έκθεση Grosset. Ρόντα. Yeah, sorry. Sorry, Chair. I'm here. Συμπαθάτε με κύριε Πρόεδρε. Εδώ κάθομαι. Εδώ, εδώ. Vi har i dag med patientdirektivet lavet Έχουμε συνάψει ιστορική σημασία συμβιβασμό, ιστορική σημασία συμφωνία. Τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ βουλευτής. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια ιστορική σημασία συμφωνία συνήθει μεταξύ δύο κομμάτων, δύο πλευρών καλύτερα, που ήταν ε, χρόνια ολόκληρα αντίπαλια δηλαδή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και καταφέραμε να συνάψουμε μια συμφωνία που αποβαίνει όφελο των ασθενών και που τους απαλλάσσει από υπερβολικά μακροχρόνιες περίοδους αναμονής. Και υπάρχει ταυτόχρονα και οικονομικός αλλά και ιατρικός έλεγχος στα ε, τεκτενόμενα, στις υπηρεσίες προσφέρονται στους ασθενείς της <coughs> Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι οφείλουμε να συγχαρούμε τους διαπραγματευτές μας και πάνω απ' όλα να ε, ευχαριστήσουμε και όλους όσους συνέπραξαν σε αυτή την ε, επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόντε. Παρακαλώ ησυχία. Ησυχία. Όποιος απαχωρεί να αποχωρήσει ησύχως. Παρακαλώ πολύ. Και στον κατάλογο έχω τον κύριο Μαστέλλα. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα υπήρχαν πολλέ αβεβαιότητε στα θέματα όσον αφορά την προσβασιμότητα στι θεραπείε και τι αποζημιώσει επιστροφέ όσον αφορά ε, τη συνολική περίθαλψη. Η οδηγία που υιοθετήθηκε επιτρέπει τελικά σε όλου του ασθενεί να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό σε όλη την ευρωπαϊκή ε, επικράτεια να έχουν δικαιώματα όσον αφορά την περίθαλψη. Ε, αυτό ενθαρρύνει δίνει τη δυνατότητα την παροχή διασυνοριακών ε, υπηρεσιών υψηλού επίπεδου. Αν αυτό είναι αναγκαίο. Χρειαζόμαστε καλύτερε πληροφορίε, μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το περιεχόμενο των διαφόρων διατάξεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά την θεραπεία που παρέχεται ε, σε άλλο κάτω μέσα από εκείνο που είναι ασφαλισμένο ασθενή. Η παρούσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Αυτή η οδηγία θα είναι μια πολύτιμη δυνατότητα για όλου του ασθενεί τη Ευρώπη, μια δυνατότητα που βασίζεται στην ανάγκη και όχι την οικονομική δυνατότητα, στην ε, ενημερωμένη ε, επιλογή και όχι στην υποχρέωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροδρίγες έχει το λόγο. Περέλα Ροδρίγκες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ισπανική συνιστόσα του Σοσιαλιστικού Κόμματος εψήφισε υπέρ το υπόλοιπο κόμμα. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι προβληματίζομαι διότι αυτή η οδηγία θίγει το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είπαμε ότι έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ με το Συμβούλιο να καλυφθεί η υπόθεση αυτή για την οδηγία. Και είδαμε αυτή στην Ολομέλεια ότι και με τις μεταμοσχεύσεις αλλά και σε άλλα νομοθετήματα εμείς θέλουμε να μην καπελωθεί με αυτό το νομοθέτημα το έργο διαφόρων φορέων όπως και του Ισπανικού φορέα ε, για την προστασία των ασθενών που έχουν υποστεί μεταμόσχευση. Οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την μεταφορά, την υλοποίηση της οδηγίας για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ κύριος Μέσσερ Σμιτ. Πρόεδρε, έχουμε εδώ να κάνουμε μια υπόθεση την οποία ε, οφείλουμε σε μια σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ε, πίεσαν ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση της οδηγίας σήμερα. Άρα θα συμφωνήσω ότι πρέπει να προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες για τους ε, Ευρωπαίους ασθενείς για περίθαλψη στο εξωτερικό. Πριν όμως με την οδηγία ε, προσφέρεται μία σημαντική ευκαιρία και πολλά πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν. Υπάρχουν χώρες, παραδείγματι, που γνωρίζουν ε, ε, δυσβάστακτους καταλόγους αναμονής ασθενών και έτσι θα μπορούσαν αυτοί να ε, εξασφαλίσουν περίθαλψη σε ένα γειτονικό κράτος. Τη Γερμανία, την Ολλανδία Φερρυπίν για ένα κράτος όπως το δικό μου η κατάσταση είναι πια αφόρητη. Και ενώ ο ασθενής πληρώνει βέβαια ως πολίτης το φόρο προς το κράτος για να έχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καταλήγει τελικά να μην την εξασφαλίζει. Αυτά λοιπόν όλα τα πλεονεκτήματα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χίγγινς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο κύριος Μέσερ Σμιτ, όντως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε με την στάση του, με την ομολογία του αυτή την ε, ε, νομοθεστική τροποποίηση, αλλά οφείλουμε μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Γκροστέτ που κατάφερε το συμβιβασμό αυτό και πρέπει να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ότι δηλαδή θα μπορέσουν πάνω από όλα ασθενείς που έχουν σπάνιες ασθένειες, εφόσον υπάρχει ε, δυνατότητα θεραπεία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, να το εξασφαλίσουν, να την εξασφαλίσουν θεραπεία εκεί. Ε, και ω εκ τούτου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση το βέλτιστο συμφέρον του ασθενούς και όχι με βάση κάποιες πιέσεις ε, και συνθήκες ε, δυσβάστακτες. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε και να αποτρέψουμε θα ήταν ο ιατρικός τουρισμός. Η ε, συμφωνία που έχει επιτευχθεί νομίζω εξασφαλίζει το πολύ θετικό της κάλυψης των αναγκών των ασθενών χωρίς όμως και να επιτρέπει τον ιατρικό τουρισμό. Μεγάλη μέρα λοιπόν για την Ευρώπη η σημερινή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και εγώ η κυρία Λουκρυπ, θέλω να χαιρετήσω τη συμφωνία της κυρίας Γκροστέτ για τη δυνατότητα πρόσβασης στις περσινοριακές ε, υπηρεσίες περίθαλψης, οτροφομακευτικής περίθαλψης και ιδιαίτερα στη δυνατότητα κινητικότητας των ασθενών από την Ευρώπη. Ύστερα από χρόνια αβεβαιότητας και πάνω απ' όλα αβεβαιότητας νομικής, δικαίου δηλαδή, και ύστερα από πολλές προσπάθειες και επίπονους ε, κόπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε με το κείμενο αυτό να διευκρινίσουμε, να κωδικοποιήσουμε και να ε, προσδιορίσουμε τους όρους από τους οποίους μπορεί ένας ασθενής να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθελψη σε νοσοκομεία του εξωτερικού, όχι μόνο προς την πρόσβαση σε αυτά τα νοσοκομεία, αλλά και ως προς την αποζημίωση των όποιων δαπανών του. Και αυτό ιδιαίτερο αποβαίνει εις όφελος των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες ασθενείς, οι οποίοι έτσι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικές, κατάλληλες και πρόσφορες για την αντιμετώπιση του, ιατρικού, του, προβλήματος υγείας από το οποίο πάσχουν. Αποβαίνει λοιπόν εις και προσφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική δε ενίσχυση και κίνητρο κινητικότητας για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Βίλαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση Γκροστέτ Ελπίζω να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το αποτέλεσμα αυτών των ε, μακροπρόθεσμων διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, ε, διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασθενών και ταυτόχρονα προασπίζει και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Για χώρε όπω η Πολωνία, η θεραπεία στο εξωτερικό σημαίνει ότι υπάρχει και ισότιμη πρόσβαση σε δυνατότητε θεραπεία. Υπάρχουν ε, μεγάλε λίστε αναμολή για δύσκολε ασθένειε και κάποιοι ασθενεί δεν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία ε, γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε κάποιες περιπτώσεις. Η δυνατότητα λοιπόν οι ασθενείς να επιλέγουν πού θα εγχειριστούν ε, ή κατά πόσον θα παραμείνουν στη χώρα τους και θα περιμένουν για την ε, θεραπεία τους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα ελπίζουμε να μπορούν να αποζημιώνονται και οι δαπάνες για αυτές τις επεμβάσεις σε όλη την Ευρώπη. Ε, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τμήμα του πακέτου της εσωτερικής αγοράς για τις ιατρικές υπηρεσίες, θα βοηθήσει στον θεμικό, το ανταγωνισμό μεταξύ των ε, υπηρεσιών υγείας και θα βελτιώσει ε, την κατάσταση για τους ασθενείς. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο ομιλίας γιατί έχουμε αρκετές επεξηγήσεις. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι καλωσορίζω και εγώ αυτή την οδηγία για την ε, υπηρεσία υγεία, αλλά ε, είμαι πολύ επιφυλακτική γιατί ο διάβολο σίγουρα θα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ε, βέβαια, η οδηγία αυτή θα τεθεί σε ισχύ σε 13 μήνε. Στο μεταξύ, βέβαια, οι ασθενεί μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα για να νοσηλευτούν στο εξωτερικό και να αποζημιωθούν για τα έξοδά του για αυτή την νοσηλεία. Να μην υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν ασθενεί οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να λοσιλευθούν και ε, ε, σίγουρα υφίσταται το θέμα. Στην ιστοσελίδα μου υπάρχει μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων ε, για το θέμα αυτό και ζητώ από τους πολίτες να μπορέσουν να ε, παρακολουθήσουν το θέμα και αν δεν έχω θέσει τις σωστές ερωτήσεις να μου το πούν διότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα γι' αυτό το νέο θετικό βήμα για την διαμεθοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι κινούνται όλο και περισσότερο, διότι ταξιδεύουμε, εργαζόμαστε και χρειαζόμαστε γιατρική περίθαλψη πέραν των συνόρων μας. Και όλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να νοσηλευτούν αν χρειαστεί σε κάποια άλλη χώρα. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να αποτρέψουμε τον ιατρικό τουρισμό, αλλά συγχρόνως θα πρέπει οι ασθενείς που χρειάζονται μια θεραπεία στο εξωτερικό να μπορούν να την έχουν. Σκέφτομαι ιδιαίτερο όλους όσους πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά κέντρα κατάστασης την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι κάνουν και τα εθνικά συστήματα υγείας στις διάφορες χώρες και πώς αντιμετωπίζουν σωστά το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιατρινάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ευρωπαϊκά μέτρα που να εξασφαλίζουν ε, ασφάλεια ιατρική, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης. Και αυτό είναι πάνω απ' όλα σημαντικό διότι ε, ρυθμίστε με μια αυτόνομη οδηγία και δεν ενσωματώθηκε στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ ελλείψει σε αυτήν την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Τα δικαιώματα λοιπόν των ασθενών. Μα δείχνει το κείμενο ότι υποχρεούνται πλέον τα κράτη-μέλη να ε, αντιμετωπίσουν ε, το πρόβλημα της μακροχρόνιας αναμονής ε, των ασθενών στο εσωτερικό τους και τα, ε, το κόστος των παροχών αυτών. Αυτό θα προκύψει ως συνέπεια της οδηγίας. Και πάνω απ' όλα η δυνατότητα για ε, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικές εκτός ε, της χώρας του ενδιαφερομένου δεν θα στηρίζεται μόνο σε οικονομικά κριτήρια αλλά και σε ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όλοι με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε σήμερα, διότι βλέπουμε ότι θα προσφέρεται ε, θα προσφέρονται υπηρεσίες υγείας, ε, η φαρμακευτική περίθαλψη στους ασθενείς ανά τον κόσμο. Ξέρετε βέβαια ότι από τη δική σας ε, περιοχή, από την Νότια Αγγλία, υπάρχουν αμφισβητήσεις και προσφυγές κατά του ε, συστήματος υγείας της Αγγλίας για τι καθυστερήσει και τα προβλήματα που παρουσιάζει. Πρέπει λοιπόν αυτό να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες μας. Αυτή είναι η δουλειά και το καθήκον του Κοινοβουλίου να συμβάλλει στις ουσιαστικέ υπηρεσίες υγείας. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε μια, ένα τρόπο ρύθμιση τη αναγνώρισης και των νεατροϊκών συνταγών, των φαρμακευτικών συνταγών δηλαδή και του τρόπου συνταγολόγηση για του ασθενεί ανά την Ευρώπη, αλλά έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Και ταυτόχρονα υπεγραμμίζω, Πρόεδρε, ότι όταν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα και μια μεγάλη οικονομική κρίση που σοβεί ανά την Ευρώπη, πολλοί είναι οι πολίτε που λένε Υπάρχει Ευρώπη, κάνει καμιά δουλειά η Ευρώπη. Και να που σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη κάνει δουλειά και καλή. Ευχαριστώ. Κύριο Μπάτεν. Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα αυτή την οδηγία για υπερσυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί θα σήμαινε αποκλειστικά και μόνο επιπλέον επιβάρυνση του, του Βρετανικού συστήματος υγείας ε, με επιπλέον άτομα που θα καταφέρουν σε αυτό και επιπλέον κόστος. Ήδη έχουμε εκατοντάδες, αν όχι δισεκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια λίρες κόστος και αυτοί που υποφέρουν περισσότερο είναι οι δικοί μου ψηφοφόροι, στο Λονδίνο δηλαδή. Άρα εδώ θα δινόταν η ευκαιρία, εάν εφόσον περνάει αυτή η οδηγία και γι' αυτό την καταψήφισα, σε οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη να έρχεται στην Ευρώπη, στη Βρετανία, να εξασφαλίζει την φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να πληρώσει δεκάρα. Είναι βέβαια σωστό να προσφέρεται κατεπίγουσα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κατάσταση ανάγκη, εφόσον είναι απαραίτητο. Αλλά όχι εάν ε, ένα τέτοιο ασθενή δεν έχει ε, προσπογράψει την κατάλληλη ασφάλιση υγεία και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ε, ήδη πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για τη Βρετανία. Αυτό είναι ακόμη ένα λόγο, η οδηγία αυτή που πέρασε δηλαδή, είναι ακόμα ένα λόγο για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Στάκκουλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό το στάδιο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, ο συμβασμός δηλαδή μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δυνατότητα ε, να αναλυφθεί δράση, να προσφερθούν αυτές οι υπηρεσίες υπερσυνοριακά. Είναι πολλές ε, οι ατελείωτες ουρές σε ορισμένα κράτη-μέλη και η χρόνια αναμονής ε, μακρύ Άρα αυτά όλα θα περικοπούν πιστεύουμε χάρη στη νέα οδηγία και πάνω απ' όλα γιατί αυτή είναι η κύρια προτεραιότητα θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια για τον πολίτη. Θα γνωρίζει τι ε, μπορεί να κάνει. Χαίρομαι ιδιαίτερως λοιπόν για την έγκριση της ε, πρότασης Γκροστέτ, της έκθεσης Γκροστέτ και ελπίζω ότι αυτή θα οδηγήσει υψηλότερο ε, βιωτικό επίπεδο, ποιότητα ζωής και πάνω απ' όλα η ιατροφαρμακευτική ασφάλεια για τον πολίτη της Ευρώπης και πέρα από τα σύνορά του ακόμα. Ευχαριστώ κύριο Ρούμπιχ. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω τα εθνικά ε, φορολογικά συστήματα να μην αποβούν εις βάρος της εσωτερικής αγοράς και στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται να έχουμε ίση μεταχείριση. Ήδη βλέπουμε κάποιο αρνητικό παράδειγμα από την ε, Ουγγαρία η οποία ε, προβαίνει σε διαφορετική φορολόγηση ορισμένων προϊόντων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Ελπίζω το ίδιο πράγμα να μην το δούμε να εμφανίζεται στο θέμα το ίση τροφαρμακευτική περίθαλψη. Και παρακαλώ τον Πρωθυπουργό Όρμπα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά αντιβαίνει στου όρου τη ελεύθερη αγορά, τη ιστορική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά. Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε. Νομίζω ότι συνολικά ένα από τα θέματα στα οποία συμφωνούμε εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ότι πιστεύουμε σε μια ε, αγαστή λειτουργία της ενίας αγοράς. Εάν λοιπόν κάποιος μου πει ότι δεν έχω καλέ υπηρεσίε στην περιφέρειά μου και θα ήθελα να ταξιδέψω στο εξωτερικό για να λάβω καλύτερα, ε, καλύτερη περίθαλψη, ε, δεν είναι βέβαιη η κατάσταση στη χώρα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι ευπρόσδεκτη η ψήφιση αυτή τη πρόταση. Θέλουμε να δούμε ε, στις περιφέρειες όπου οι ασθενεί δεν λαμβάνουν καλή περίθαλψη να μπορούν μέσω αυτή τη οδηγία να περάσουν σε μια άλλη χώρα μέλο, πιέζοντας έτσι και τα εθνικά συστήματα υγείας να βελτιωθούν, να βελτιώσουν τι υπηρεσίε του ώστε να ε, ανταποκρίνονται στι ανάγκε των ασθενών του. Επίση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διευκολύνουμε τη διαδικασία μέσω τη οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για το κόστο το οποίο κατέβαλαν οι ασθενεί ε, τη χώρα του ε, όταν νοσηλεύτηκαν σε άλλη χώρα. Θέλουμε να φροντίσουμε να εφαρμοστεί καταλήλω η οδηγία. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα ε, στην ε, συμφωνία, ε, θελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης για το FLEGD. Ο κύριος Higgins. Υπερψήφισα τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Καμερούν και το Κονγκό για την συμφωνία αυτή για τις χώρες θα πρέπει να διατηρηθούν τα τροπικά δάση για να υπάρχει ε, ισορροπία στα οικοσυστήματά μας και θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους αυτόχθονες πληθυσμούς ε, που ζουν στα δάση αυτά ε, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν την εκμετάλλευση του περιβάλλοντός τους, την υλοτόμηση μεγάλων εκτάσεων από επιχειρήσεις και αυτά όλα γίνονται ε, για να υπάρχει κέρδος. Ε, κατέθεσα μία τροπολογία ώστε ε, η δασική βιομηχανία να ελέγχεται δημοκρατικώς από τους εργαζόμενους και τους αυτόχθονες που ζουν στα δάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έκθεση Μάρτιν τώρα. Ο κύριος Μέσερσμιτ. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι... Αυτό είναι ο μόνο τρόπο ε, να οδεύσουμε προ την ευημερία ω ενιαία αγορά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τι χώρε οι οποίε είναι υπό ανάπτυξη. Πρόκειται για τη μόνη πρωτοβουλία ανάπτυξη την οποία μπορούμε να υπερασπιστούμε εάν ε, λάβουμε υπόψη αυτό που κάνουν ε, οι άλλες μεγάλες περιοχές ε, στον κόσμο και τι στρατηγική ακολουθούν, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι κινούνται όλο ένα και ταχύτερα. Υπάρχει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Μερκοσούρ, με τις χώρες της Ασίας και η μόνη περιοχή η οποία ακόμα είναι αποκλεισμένη και δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης είναι... Ακριβώς η περιοχή αυτή. Η περιοχή λοιπόν, ε, ε, η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με τα νησιά Φίτζι και τη Γουινέα δεν είναι και το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τόσα χρόνια κάναμε διαπραγματεύσεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία, οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν τις θέσεις μες εργασίας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέκονται στο ύψος των ε, προκλήσεων για τους πολίτες τους οι πιο ελεύθερες είναι οι πιο ευημερούσες κοινωνίες. Και συμβαίνει και το αντίθετο. Θα πρέπει βεβαίως εδώ να αναγνωρίσουμε το ρόλο που παίζει το ελεύθερο εμπόριο. Όταν πρόκειται τώρα για πολυμερείς συζητήσει για το εμπόριο, ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι αυτό ο οποίο θέτει του κανόνε και γι' αυτό έχουμε περισσότερε διμερεί συμφωνίε. Και δεν μπορούν να εποφεληθούν πάρα πολύ οι πολίτες των φτωχότερων ε, χωρών εάν δεν συνάψουν διμερείς συμφωνίες. Θα πρέπει όμως σιγά σιγά τα συμφέροντα των καταναλωτών να έχουν περισσότερο ε, υπόψη από αυτά των εμπόρων. Γιατί οι καταναλωτές με ρωτούν πολλές φορές δεν έχουν την ίδια επιλογή που έχουν και οι χώρες οι ευημερούς συστήτες Και για να καθώσουμε, να τους δώσουμε αυτό που ζητούν θα πρέπει να μπορέσουμε να ευνοήσουμε ακόμη περισσότερο το ελεύθερο εμπόριο για να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες του κόσμου. Κύριε Ντίβα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Και πολλά χρόνια η περιοχή του Ειρηνικού ήταν η σταχτοπούτα των αναπτυξιακών πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πρωτοβουλίες των Φίτζη και της Γουινέας Παπουαζίας με τις ε, εταιρικές εμπορικές σχέσεις όχι θα διευκολύνουν το ελεύθερο εμπόριο με αλλά και μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από αυτή τη συμφωνία μέχρι τώρα είναι ότι οι κανόνες προέλευσης στην Ιταλία θα επιτρέψουν τα άτομα που ζουν στην περιοχή του Ειρηνικού να βάλουν στην, κάποια προστιθέμενη αξία στην αλία τους. Είναι περιοχές που έχουν ε, πάρα πολλές ε, ε, ποσότητες αλλιεύματα. Τώρα μπορούν να εξάγουν τα αλλιεύματα τα οποία θα τα έχουν επεξεργαστεί και στις άλλες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταπολεμήσουν και την φτώχεια. Τώρα περνάμε στη Εθνή Υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα υπερψήφισα την προφορική ερώτηση για τις διεθνείς υιοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής υιοθεσία είναι η διαδικασία η οποία μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να υπάρχει μόνιμη οικογένεια για τα παιδιά για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί ιδανική οικογένεια στη χώρα καταγωγής τους. Η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών ε, στα κράτη-μέλη σε θέματα διεθνών υιοθεσιών είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η οθεσία θα γίνεται προ συμφέρον του ανηλίκου, ε, προ την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και δεν θα υπάρχει πώληση και εμπορία παιδιών. Επίση, θα πρέπει να προβλέψουμε απλούστευση τη διαδικασία διεθνών υιοθεσιών, οι οποίε πολύ συχνά ε, λόγω ε, γραφειοκρατικών προσκομμάτων ε, αποτελούν αντικίνητρο για τις οικογένειες οι οποίες θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Η περίπτωση της Ρουμανίας που είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει απαγορεύσει δια νόμου τις διεθνείς υιοθεσίες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε σήμερα 70.000 ορφανά παιδιά, τα περισσότερα βρίσκονται στα ορφανοτροφία και πολλά από αυτά βρίσκονται σε ανάδοχες οικογένειες. Θα πρέπει να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να βρεθούν σε νέες οικογένειες μέσω διεθνών υιοθεσιών. Η κυρία Σάσκοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να παραστώ στην συζήτηση την Δευτέρα λόγω της υποχρέωσης να ασχοληθώ με τα δικά μου παιδιά. Θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου στο ψήφισμα και να εκφράσω την ελπίδα η συνέχεια που θα δοθεί στο ψήφισμα αυτό να σημάνει και περιορισμό του γραφειοκρατικού φόρτου σε αυτές τις διεθνείς υιοθεσίες και πάνω απ' όλα μια καλύτερη παρακολούθηση του τι συμβαίνει στην οικογένεια μετά την υιοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως είναι πολλοί οι συνάδελφοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έναν αδυσόπιτο πόλεμο λέξεων που σοβεί εδώ στην υπόθεση της διεθνούς υιοθεσίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε τις λέξεις και να κοιτάξουμε την ουσία. Εμείς αυτό που πράξαμε ήταν να επιλέξουμε την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Και αυτό σημαίνει ότι προστατεύουμε οποιοδήποτε παιδί, οπουδήποτε και αν έχει γεννηθεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην καταφερόμαστε κατά ιουδήποτε συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι σε κάθε κράτος υπάρχουν παιδιά εγκαταλελειμμένα ή παιδιά τα οποία δεν εξασφαλίζουν την απαραίτητη στοργή και φροντίδα μέσα στην οικογένεια την οικογένεια πυρήνα όπως την γνωρίζουμε και που χρειάζεται να δοθούν σε άλλες οικογένειες. Ας μην ε, περιορίσουμε όμως πέραν αυτής της διάστασης και τη διάσταση της παρακολούθησης εφαρμογής νομοθεσίας. Και επίσης ήθελα να πω ότι υπάρχουν ε, κάποιοι γονείς οι οποίοι καταβάλουν πολύ περισσότερο κόπο και δίνουν πολύ περισσότερη αγάπη στα παιδιά από αυτούς που ονομάζονται ε, βιολογικοί εικονείς, αυτοί δηλαδή που δίνουν ε, τη ζωή στα παιδιά. Η κυρία Ροντζούλη, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή Σκέφτομαι χιλιάδες ζευγάρια που καθημερινά αντιμετωπίζουν ε, ε, δυσκολίες και προσπαθούν ε, να υιοθετήσουν ένα παιδί. Η υιοθεσία είναι αξία, είναι μια εκδήλωση αγάπης που ανοίγει τις πόρτες για μια νέα οικογένεια για ένα παιδί που δυστυχώς δεν μπορεί ακόμα να βασίζεται στη στοργή των φυσικών του γονιών. Ε, κάθε παιδί που εγκαταλείπεται έχει δικαίωμα να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ε, το οποίο θα του προσφέρει ευτυχία. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε η ηρεμία αυτή να μην αποτελεί πλέον ουτοπία. Σήμερα με την προφορική αυτή ερώτηση θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στο θέμα αυτό και να δημιουργήσουμε νέα νομοθεσία για να βελτιώσουμε αυτές τις νομοθεσίες τις υιοθεσίες. Ε, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσκομα για τα όνειρα και την επιθυμία ενός παιδιού να αποκτήσει μια νέα οικογένεια. Η κυρία Ντότς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την πρόταση ψηφίσματο ε, για τι διεθνεί υιοθεσίε ε, που ψηφίσαμε σήμερα. Γνωρίζω πάρα πολλού ανθρώπου ε, στην περιφέρειά μου που πέρασαν ή περνούν τώρα από αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά είναι ε, ανεκτήμητη η αξία του να έχει κάποιο οικογένεια και παιδιά. Αλλά το να φτάσουμε πολλέ φορέ στην υιοθεσία είναι μακρύ ο δρόμο και πολλέ διαδικασίε μπορεί να καθυστερήσουν και πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία και εμεί θα πρέπει ω Κοινοβούλιο να αναζητήσουμε αναζητήσουμε τρόπους να μειωθεί αυτή η γραφειοκρατία και να έχουμε μια πιο εξορθρολογισμένη διαδικασία. Εκ παραλίλου όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες και την ασφάλεια των παιδιών διότι πολλά από αυτά έχουν ε, μεγάλες ανάγκες και θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ώστε τα παιδιά να μην δίνονται σε οικογένειες οι οποίες μπορεί να είναι ευάλωτα όμως ελοχεύει και ο κίνδυνος ε, άνθρωποι που μπορεί να τα αγαπήσουν και να τα φροντίσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και αυτό φυσικά ε, είναι πρόβλημα για τα παιδιά. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διεθνούς υιοθεσία. Πλέον το σημερινό ψήφισμα προσπαθεί να δώσει μια όθηση σε μια ε, κατάσταση η οποία γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Η άφηξη νέων χωρών αντί να αποτελέσει κίνητρο για τις διεθνείς υιοθεσίες έχει ε, δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία και πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά και δεν μπορούν να δώσουν ευτυχία σε ένα παιδί μετά από πάρα πολλές ε, προσπάθειες στη χώρα τους. Υπάρχει όλο και περισσότερη γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει τη μειοθεσία παιδιών Ταυτόχρονα αυξάνεται και η εμπορία οργάνων και τα θέματα της προστασίας των ανηλίκων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτή την πρόταση ψηφίσματος και να δώσουμε την κατάλληλη ε, δυνατότητα να επιταχυνθούν ε, οι διαδικασίες διεθνούς υιοθεσίες και να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή υιοθεσία για να δοθεί ένα μέλλον σε τόσα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ κύριε Γκέρλινγκ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ασκεί την Προεδρία με αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ σοβαρό θέμα. Η διεθνή υιοθεσία βεβαίω είναι πρωταρχική σημασία και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Και χαιρετίζω το ψήφισμα αυτό, το οποίο λέγει πω πολλά ψηφίσματα τα οποία εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλά λογικά και ευφυή πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω πραγματικά να πω και έμαθα πολλά βοηθώντας ε, στην δική μου εκλογική περιφέρεια είναι ότι δεν είναι το θέμα το οποίο ε, είναι σημαντικό δεν είναι να προσπαθήσουμε να, σε ένα τόσο δύσκολο θέμα να ρίξουμε φως και να απλοποιήσουμε την κατάσταση και διάφορες οργανώσεις να δραστούν Θα ήθελα αυτά τα σωστά επιχειρήματα να τα κάνουμε πράξη. Δηλαδή, να απλοποιηθούν τα πράγματα, να γίνουν πιο σωστά. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κάνει τίποτα και αντί να απλοποιήσουμε την κατάσταση και να κάνουμε τα πράγματα πιο αποδοτικά, θα τα κάνουμε ακόμη πιο δύσκολα. Ευχαριστώ. κύριο Τάκουλα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την υποστήριξή μου για αυτή τη συμφωνία για τη διεθνή υιοθεσία Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τέτοιες ιστορίες ε, εκ του σύνεγγες και γνωρίζω ότι η κατάργηση της, νομοθεσ... της γραφειοκρατίας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υιοθεσίας των παιδιών αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διαφυλαχθεί πάντοτε η δεοντολογία και η ηθική δηλαδή κάθε δράση που θα αναλαμβάνεται ως προς την υιοθεσία να μην έχει σχέση με εμπόριο παιδιών δεν μπορούμε να βλέπουμε το παιδί ως ένα ε, αντικείμενο αλλά ως έναν άνθρωπο, έναν ανθρώπινο όν, στο οποίο προσφέρουμε αγάπη και στοργή μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον. Και ταυτόχρονα θα πρέπει το παιδί να έχει δικαιώματα και δυνατότητα να χαρεί την αγάπη και τη στοργή ενός πατέρα και μιας μητέρας. Αυτός πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας και ο τελικός μας στόχος. Δεν είναι όμως πάντα αυτά τα πράγματα απλά. Υπάρχουν και πολιτισμικές διαφορές. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μερικές φορές αντικατοπτρίζονται και στο DNA του καθενός μας. Αλλά πάντως πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε στο παιδί αυτό που υιοθετούμε μια ισορροπημένη οικογένεια και ε, υποδοχή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Σερβίας, ο κύριος Μέσερ Σμιτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η χώρα που βασανίστηκε περισσότερο τα περισσότερα χίλια με δύο χρόνια είναι η Σερβία. Οι Γερμανοί, οι Ρώσοι πέρασαν από εκεί. Και σήμερα έχουμε την δυνατότητα να αναστρέψουμε την κατάσταση νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ελπίδες για τη χώρα αυτή. Ξέρουμε ότι πριν από μερικά χρόνια το ΝΑΤΟ κατέστρεψε τη χώρα αυτή, την πρωτεύουσά της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε πολλά πράγματα. Ξέρουμε τι έγινε επίσης στο Κωσυφοπαίδιο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει σήμερα να ξεχάσουμε τι έγινε στο παρελθόν, να κοιτάξουμε το μέλλον και να δούμε αυτή την φίλη χώρα και να την ε, βοηθήσουμε να προχωρήσει. Ο κύριος Νικολάς. Η συμφωνία αυτή σταθεροποίηση και σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σερβία θα δημιουργήσει βάση για στενέ σχέσει βάσει της αμοιβαιότητας και των κοινών συμφερόντων και θα προσφέρει στην περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Είναι μοναδική ευκαιρία να αλλάξει η χώρα, να γίνει πιο ευημερής, να εξυγχρονιστεί η οικονομία της και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να βελτιώσει την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την δημόσια διοίκησή της, να εφαρμόσει σωστά τις αρχές της δικαιοσύνης και να βελτιώσει το σύστημα το δικαιοσύνης και το δικαστικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν θέματα κατά στρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να έχει και στενή συνεργασία με το ε, δικαστήριο της Χάγης της Σερβίας. Ευχαριστώ κύριος Καλανάσκη. Στην επόμενη έκθεση θα ήθελα να λάβω το λόγο κυρία Πρόεδρε. την έκθεση Ματιάς. Το σημειώνουμε. Ο κύριος Χάνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας και τους διερμηνείς για την ε, υπομονή σας. Βασισμένη στην επιλογή μεταξύ υπερεθνικισμού και δημοκρατίας, εμείς είμαστε πάντα ε, δημοκρατία. της δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει στα Βαλκάνια. Σε πολλές χώρες, την ε, Βοσνία, στην ε, Μακεδονία και σε άλλες χώρες, ο καθένας προσπαθεί να διασφαλίσει τα εθνικά του σύνορα και είναι δύσκολο να έχει κανείς μία δημοκρατία που να λειτουργεί εάν δεν αισθάνονται ένα κοινό αίσθημα οι λαοί μεταξύ τους και οι κυβερνήσεις τους. Διότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να αναγνωρίζει παρά το ότι αναγνωρίζει την ε, ταυτότητά του και κάποιες εθνικές αρχές και τους άλλους. Για να υπάρχει δημοκρατία πρέπει να υπάρχει δήμος. Και νομίζω ότι εάν αφαιρέσει κανείς ε, τον Δήμο από την δημοκρατία δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει μια σωστή λειτουργία χώρα. Ευχαριστώ κύριο Στίβ. Uh, you have a problem with your microphone again. Yes, I do, yes. Έχετε πρόβλημα με το μικρόφωνο σας. Πολύ καλά νέα, κυρία Πρόεδρε. Όταν υπενθυμίζουμε, όταν θυμόμαστε από πόσο μακριά έρχεται η Σερβία στα πλαίσια του Εθνούς Δικαίου και του κράτους δικαίου, εάν δούμε πώς ήταν η Σερβία πριν από 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα, θα πρέπει να επενέσουμε την ε, δίκη στη Σερβία για τα βήματα που έκανε. Διότι μπόρεσε να γίνει σιγά σιγά η χώρα ένα κράτος δικαίου. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό το Υπάρχει συνεργαστία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού ε, συστήματος επίσης γίνονται και βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές. Είναι λοιπόν μεγάλα τα επιτέματα και τα κριτήρια της Κοπενχάγης νομίζω ότι πληρούνται σιγά σιγά. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία αντιμετώπισε ένα πάρα πολύ δύσκολο πόλεμο και σήμερα αναδύεται σαν μια χώρα η οποία θα είναι καλός εταίρος και με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό είμαι υπέρ της Συμφωνίας Συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Έκθεση Κατσίν. Κύριος Μπίλαν, παρακαλώ. Πρόεδρε, το δικό μου, η δική μου παρέμβαση έχει να κάνει με την Σερβία, υπεξήγηση ψήφου. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας αποτελεί ορόσημο στο δρόμο που έχει πάρει αυτή η χώρα στην ένταξη με την στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την υποστηρίξουμε σε κάθε της βήμα. Υποστηρίζω λοιπόν τη ε, συμφωνία αυτή και καλό και τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν το ταχύτερο δυνατό. η στενότερη συνεργασία τη ε, Σερβία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημάνει ταυτόχρονα και στενότερη ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, Εγκλημάτων Πολέμου τη Χάγη και αντιμετώπιση πιο ουσιαστική των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μειονότητα των Ρωμά. Ιδιαίτερα όμως χαιρετίζω την έμφαση που δίνεται στη δημοκρατία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες που συνάπτονται. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάμε στην έκθεση της και τον κύριο μας Στέλλα πρώτα-πρώτα. Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας ε, είναι πολύ σημαντικές ε, και σας το λέω γιατί και ο πατέρας μου έπασχε από Αλσχάιμερ και η γιαγιά μου. Ελπίζω να είμαι εγώ στο τέλος αυτού του γενετικού κρίκου. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι κατάλληλες ε, ε, ιατρικές φροντίδες στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νόσους. Θα πρέπει να υπάρχει καταπολέμηση των διαφορών που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο και να μην υπάρχει και ανοσότητα στη διαδικασία περίθαλψης. Θα πρέπει να προάγουμε την πρόληψη και την ποιότητα ζωής και να βελτιώσουμε τις γνώσεις, την παθολογία και να συντονίσουμε και τις έρευνες οι οποίες είναι εξελίξη να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των, κρατών μελών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Με την παρούσα έκθεση ζητάμε επίση και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια απάντηση πιο συντονισμένη για την πρόληψη, την ε, ε, θεραπεία ε, των ε, διαφόρων μορφών της άνοιας, κυρίως του Αλσχάιμερ και για όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας αλλά και για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Και θα μπορέσουμε να έχουμε συνένεση μόνο με την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν προτεραιότητα για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε υπερψήφισα αυτή την έκθεση και χαίρομαι που πέρασε η έκθεση. Πήγα σε όλε τι συζητήσει στο Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώ δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μέχρι τούδε. Επομένω, εκμεταλλεύομαι τη δυνατότητα που μου δίνεται εδώ για να αναφέρω κάποια σημαντικά στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζεται κατάλληλα έρευνα για να μπορέσουμε να ζητήσουμε τα αίτια αυτή τη νόσου. τι ρόλο διαδραματίζουν ε, οι διάφοροι παράγοντες όπως για παράδειγμα η γενετική στην ε, εμφάνιση της νόσου γιατί είναι περισσότερες οι γυναίκες που νοσούν σε σχέση με τους άνδρες και αυτά όλα τα ερωτήματα είναι δύσκολα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε και ε, ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι η έρευνα. Πρέπει να υπάρξει έρευνα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια θεραπεία για την νόσο και να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριο Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η νόσος του Αλσχάιμερ είναι μία εξ αυτών για τις οποίες δεν διαθέτουμε ακόμα θεραπεία. Και επειδή έχουμε όλο και περισσότερο, ε, ε, ε, περισσότερο γυράσκων πληθυσμό θα έχουμε ακόμα, περισσότερες και, ε, ακόμα περισσότερα περιστακτικά. Η άνοια δεν αφορά μόνο όσους πλήττονται από αυτήν αλλά και όσους του φροντίζουν και το οικογενειακό τους και φιλικό τους περιβάλλον. Η έκθεση αυτή επισημαίνει που έγινε τα προβλήματα και προσπαθεί να βελτιώσει και την περίθαλψη. τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάλληλα σχέδια για να βοηθήσουν και τους ασθενείς αλλά και όσους τους περιβάλλουν και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε προκειμένου να μειωθούν οι ασθενείς και τα άτομα τα οποία πάσχουν από την νόσο ε, ε, στο μέλλον. Οι πνευστήρες για ασθηματικούς. Τώρα, ο κύριος Χίγκιν. Είχα ζητήσει και χρόνο αγόρευσης ε, για την ε, προηγούμενη έκθεση, για, την για το αλσχάιμερ, αν μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αντιμετωπίζει από πολλές πτυχές το εφαλτήριο για την νόσο του Αλσχάιμερ. Μιλάμε για την πρόληψη, μιλάμε για την ε, θεραπεία και για την αντιμετώπιση. ο άνθρωπος φοβάται διάφορες ασθένειες και η μεγαλύτεροι φόβη είναι για το Αλσχάιμερ και τον καρκίνο. Καταρχήν πρέπει να διαγνώσουμε τα αίτια του καρκίνου, την πρόληψη του από εκεί και πέρα και να δούμε τι θα γίνει και από πλευρά θεραπεία. Στον καρκίνο έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ε, παρά το γεγονό ότι η νόσος του Αλσχάιμερ ε, ε, ανακαλύφθηκε το 1906 και ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με την ε, άνοια, ε, δεν ξέρουμε τι το προκαλεί και δεν ξέρουμε ακόμα πώς να τη θεραπεύσουμε. Οι μεγάλες προκλήσεις όμως είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, να ε, ε, βρούμε ποια είναι τα αίτια και να προλαμβάνουμε και να καταλήξουμε και σε μια θεραπεία. Ευχαριστώ να υποθέσω κύριε Χίγγινς ότι δεν θέλετε να μιλήσετε για τους εισπνευστήρες, για τους ασθηματικούς. Η κυρία Μάτερα και η κυρία Μουσκαρδίνη είχαν ζητήσει το λόγο, αλλά έχουν φύγει από την αίθουσα. Επομένως θα προχωρήσουμε τώρα στην κατάσταση στην ΑΕΤ. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσοι έχουν επισκεφθεί την ΑΕΤ είδαν τις μεγάλες ε, κατασκοφές και βλέπουμε, είδαμε τι συμβαίνει και σωστό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι κοινοτικοί όλοι οι οργανισμοί για βοήθεια έφεσαν τις δυνάμει από κοινού για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Σήμερα όμως θα πρέπει να δούμε την κατάσταση ένα χρόνο μετά. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα τα οποία τονίζονται εδώ σε ψήφισμα Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μεγάλα προβλήματα ε, υγείας ακόμη, προβλήματα στεγαστικά και γίνεται ε, η Επιτροπή σε συνεργασία με τη ΔΕΦ κυβέρνηση έχει κάτι βάλει πάρα πολλέ προσπάθειε, αλλά κάτι το οποίο λείπει είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα. Εάν μακροπρόθεσμα πρέπει, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα βραχυπρόθεσμα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, θα πρέπει ο ιδιωτικό τομέα εμπράκτο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι για να βοηθήσει. Ο κύριο Δίβα. 5% της ε, ε, λάσπης ε, έχει 230,000 are dead, 300,000 Ότι έχει μείνει από τα γκρεμισμένα κτίρια έχει μόνον μπορέσει να μαζευτεί. Για ποιο λόγο. Γιατί μόνο 5% έχει καθιστεί. Όταν έχετε έναν σεισμό Πρέπει να υπάρχουν μηχανήματα που θα καθαρίσουν. Ποιο θα μπορέσει εκεί πέρα, με φτιάρια ή μη κυβερνητικέ οργανώσει. Αυτό το οποίο αυτό μόνο μπορούν να το κάνουν αποτελεσματικά ε, αυτοί που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, βαρύ εξοπλισμό. Ο στρατός. Και τι συμβαίνει. Εάν δεν μπορεί να βοηθήσει ε, θέλει να βοηθήσει ο στρατό, αλλά η άκρα αριστερά και του Κοινοβουλίου και αλλού λέει να σηκωθούν να φύγουν. Έτσι λοιπόν τα πράγματα εδώ και ένα χρόνο παραμένουν ως ήταν. Αυτό λοιπόν από πολιτικής απόψεω είναι λανθασμένο. Δηλαδή κανείς να μην μπορεί να καταλάβει και ιδιαίτερα η αριστερά του Κοινοβουλίου ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι ντροπή για την παγκόσμια κοινότητα. Τώρα. Στο επόμενο θέμα, παραβίαση τη ελευθερία έκφραση και διακρίση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία. Κύριε Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως προς την κατάσταση στην ΡΑΙΤΗ. Επιτρέψτε μου δύο λόγια. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι υπήρξαν προβλήματα στον συντονισμό της βοήθειας. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό για να επιταχυνθεί και η αντιμετώπιση των συνεπειών ε, του σεισμού και η παροχή βοήθειας. Το ανέφερε και ο κύριος Δέβα τώρα, αλλά δεν μπορεί αυτό να το προσφέρει κανείς μεμονωμένα. Χρειάζεται ολόκληρη η κοινότητα, ολόκληρη η κοινωνία να δώσουν τη στήριξή τους κατά τρόπο συντονισμένο. Και όντως, δυστυχώς, Οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι δεν έγιναν πολλά στην ΑΕΤ. Πολλέ ήταν χριστιανικέ οργανώσει που αγωνίζονται, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για να βελτιώσουν έστω την καθημερινή ζωή αυτών των ανθρώπων στην ΑΕΤ και πρέπει να τις τιμήσουμε και να τις στηρίξουμε. Πλην όμω χρειάζεται καλύτερο συντονισμό τη παρουσίας τη Ευρώπη και των μέτρων που λαμβάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Α πάμε τώρα στη Λιθουανία. Ο κύριος Φαντάλε. Κύριε Πρόεδρε, η Λιθουανία προτείνει μέσα από το κοινοβούλιο της μια νέα σειρά προτάσεων για τους ε, και τις ομοφιλοφίλους. Έχουμε να κάνουμε μια χώρα που λειτουργεί, όπου λειτουργεί ικανοποιητικά η δημοκρατία, όπου όμως δύο φορές ο πρόεδρος της χώρας ανέπεμψε το κείμενο, το απέρριψε δηλαδή. Είναι δύσκολο να δούμε τι έκβαση θα έχουν συστήσει. Οι νέε συστήσει πρόκειται να γίνουν στο Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να δώσει κάποιες ηθικές κατευθύνσεις για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ε, επιβληθεί με τη νέα νομοθεσία στη Λουθόνια. Αλλά εάν πρόκειται να επιβληθεί νέα νομοθεσία, α δούμε πρώτα απ' όλα τι θα, τι θα περιέχει και τι θα προβλέπει. Αλλά μιλισμονούμε ταυτόχρονα ότι την πρώτη και την τελευταία λέξη την έχουν οι βουλευτέ τη χώρα. Προσωπικά το κείμενο που προτείνεται μου φαίνεται απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικολάσιτσκ. Πρόεδρε. την έγκριση εσωτερικής νομοθεσίας την αναγνωρίζουμε μόνο ω αρμοδιότητα αποκλειστική του Εθνικού Κοινοβουλίου. Έτσι συμβαίνει και στην Λιθουανία. Καλό λοιπόν θα είναι πάντοτε να θυμούμαστε ότι το θέμα των σεξουαλικών δικαιωμάτων υπάγεται στην οικογενειακή νομοθεσία, στην νομοθεσία για την οικογένεια ενό κράτου μέλου, δηλαδή ανοίξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτου μέλου. Έχει την αρμοδιότητα η πολιτεία κάθε χώρας να ορίζει και ποια είναι τα δικαιώματα και ποιος είναι ο τρόπος προστασίας των παιδιών στη χώρα αυτή και με ποιες συνθήκες θα ε, λειτουργεί ε, η νομοθεσία σχετικά με την, σχετική με την νομοθεσία. Η προστασία λοιπόν των παιδιών από βλαπτική για αυτά νομοθεσία από νομοθεσία που μπορεί αρνητικά να επηρεάσει την ε, ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός παιδιού είναι αποκλειστική αρμοδιότητας του κράτους μέλους. Μόνο αυτό μπορεί να κρίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό για ένα παιδί. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λάντσπερκης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τα σχόλιά μου για το ε, ψήφισμα που καταδικάζει την Λιθουανία. Είναι τα εξής, ότι δεν λαμβάνει υπόψη το πιο σημαντικό σημείο το κείμενο αυτό και ήθελα αλλά δεν κατάφερα να ε, συμπεριλάβω στο κείμενο ε, μία προφορική τροπολογία πολύ σημαντική κατά την άποψή μου ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίκειται στις βασικές αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της επικουρικότητας για τα κράτη-μέλη να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και να σχολιάζει ή να ζητεί τροποποίηση εθνική νομοθεσία. Αυτό δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το κάνει γιατί υπενθυμίζει παλιέ σοβιετικέ, τακτικέ και τα υπόλοιπα στο κείμενο συνεχίζουν όπω είχε. Και συνεχίζω ακόμη με μια άλλη προφορική τροπολογία ότι το πρόσχημα για τέτοιο ψήφισμα ξεκίνησε από ένα σχέδιο τροπολογίας που είχε ε, υποβάλλει μόνο ένα μεμονωμένο βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλίου. Το υπογραμμίζω. Ένα μεμονωμένο βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλίου και παρόλα αυτά στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τρόπο επίμονο, παράλογο, ε, αναφέρεται στον πληθυντικό ε, ο όρο βουλευτέ, μόνο και μόνο για να δοθεί εντύπωση και μάλιστα έξι φορέ ότι υπάρχουν πολλαπλέ τροπολογίε και, παρεμβα... και ε, τέτοιες προσπάθειες βουλευτών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε... Κύριε Λαντσπέργκη, παρακαλώ τέλειω το λεπτό σα. Όχι Πρόεδρε, εδώ έχουμε να κάνουμε μία πρόταση ενό μόνο βουλευτού και όχι απόφαση ενό Ευρω... Εθνικού Κοινοβουλίου που κατηγορείται τελικά με αυτό το ψήφισμα πώ παραβιάζει του κανόνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Είναι αυτό ο παραλογισμός του, της σύνταξης των κειμένων ασχέτως και της ευθύνης για την υποβολή προτάσεων και κειμένων που έχουμε συντάξει τα οποία θα έπρεπε ή μη τι άλλο να έχουν στηριχθεί σε κάποια ευφυή συνεργασία και να μην πρόκειται για σκύβαλα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο είναι ο κύριο Χάνων και παρακαλώ αφήστε μα να πάμε για φαΐ επιτέλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και δεκαετίε τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τον νόμο, την ισότητα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα οπισθοδρόμηση σε καμία χώρα ε, και καμία διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Πρόκειται για πρόταση, όπως είπε ο συνάδελφος. Δεν πρόκειται για νομοθετικό ψήφισμα. Αν θυμάστε, και εμεί στη Μεγάλη Βρετανία είχαμε τέτοιου είδους συζητήσεις και επιχειρήματα. Εγώ ήμουν κατά ακόμη και του δικού μου ε, κόμματο στην αρχή, διότι μου φαίνεται ότι είναι απαράδεκτο ο νόμος να ε, χρησιμοποιείται ω μέσον για να κάνουμε κάποια διάκριση αρνητική θετική για κάποιον. Εγώ όμω δεν είμαι νομοθέτη στην Λιθουανία. Μπορεί ο καθένα να έχει τι απόψει του εδώ για την έκτρο, για το οτιδήποτε, για το τι συμβαίνει σε άλλε χώρε, για την μία χώρα από την άλλη. Αλλά πρόκειται για θέματα τα οποία πρέπει να ε, τα χειρίζεται ο κάθε εθνικό νομοθέτη και κάθε χώρα και να αναγνωρίζει και πρέπει εμεί όλοι να αναγνωρίσουμε το κυρίαρχο δικαίωμα που έχει κάθε χώρα να κάνει τους δικούς της νόμους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, έληξε η συνεδρίαση. Θα επανέλθουμε στις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς που υπομονετικά εργάστηκαν ως τώρα.